Possiamo Ας ξεκινήσουμε τις εργασίες μας. Καλησπέρα σε όλους. Έχουμε πολλά θέματα στη σημερινή ημερήσια διάταξη και πολλές ψηφοφορίες. Ας ξεκινήσουμε όμως με κάποιες ανακοινώσεις. Μαγνητοσκοπείται η σημερινή μα συνεδρίαση και μεταδίδεται σε ζωντανή μετάδοση μέσω του διαδικτύου. Σας έχει δοθεί ήδη από τι 3 Οκτωβρίου το σχέδιο μερίσιας διάταξης και στις 9 Οκτωβρίου η Επιτροπή Προπολογισμών ενέκρινε μια έκθεση για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο στις 10 Οκτωβρίου η διάσκεψη των Προέδρων ενέγραψε το σημείο αυτό στην δεύτερη ολομέλεια του Οκτωβρίου. Τότε λοιπόν θα γίνει η ψηφοφορία. Πράγμα το οποίο ότι εμεί σήμερα θα πρέπει να ψηφίσουμε τη δική μας την γνωμοδότηση, την έκθεση Τρασκόφσκι. Ξέρετε ότι έχουμε δύο πολύ σημαντικές εκθέσεις από θεσμικής πλευράς σημαντικές, οι οποίες ε, θα ψηφιστούν στην Ολομέλεια του Νοεμβρίου. Καθώ επίση και δύο γνωμοδοτήσει οι οποίε θα πρέπει να διαβαστούν στι καθήλυνα αρμόδιε επιτροπέ. Αν δεν έχετε λοιπόν αντιρρήσει, μπορούμε να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Τώρα, όσον αφορά τι ανακοινώσει του Προέδρου, σημείο 2. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα μα ενημέρωσε ότι η αντιπροεδρό μα, η κυρία Κωνσταντ Λεγκρίπ, θα είναι η συγγήτρια για τον ενιαίο μηχανισμό εξυγίανση για την Τραπεζική Ένωση. και ο κύριος Μάρτι θα είναι ο εισηγητής για τον κανονισμό 90 όσον αφορά τον, α, τις διεθνείς συμφωνίες. Οι αποφάσεις αυτές ελήφθησαν στην τελευταία μας συνεδρίαση. Αν, δεν υπάρχουν λοιπόν αντιρρήσεις μπορούμε να θεωρήσουμε ότι εγκρίνεται η πρόταση αυτή και αυτός ο διορισμός εισηγητών. Πρέπει να σας πω επίσης ότι τα διάφορα έγγραφα της ε, συνεδρίασής μας ε, είναι διαθέσιμα πλέον και ηλεκτρονικά μέσω email, μέσω του ε, e-meeting. Αλλά βέβαια θα λαμβάνετε και τα έγγραφα αυτά σε έντυπη μορφή. Πρέπει να σας πω επίσης ότι στις 26 Νοεμβρίου, την 3η 26 Νοεμβρίου, θα λάβει χώρα στη πλαίσια της δικής μας Επιτροπής μία έκτακτη συνεδρίαση υπό τη μορφή σεμιναρίου, προκειμένου να καταφέρουμε να αρχίσουμε να εφαρμόζουμε το άρθρο 17 της Συνθήκης της Λισαβόνας, όπου προβλέπεται ότι μπορούν να συμβάλλουν στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και οι εκκλησίες, οι θρησκευτικές οργανώσεις και κοινότητες, οι φιλοσοφικές και μη ομολογιακές οργανώσεις. Ο αντιπρόεδρος μας λοιπόν ο κύριος ε, Λάσλο Σούριαν είναι αρμόδιος για τα ζητήματα αυτά και μαζί του αποφασίσαμε να, να διοργανωθεί μια συνεδρίαση όπου θα προεδρεύει ο υποφαινόμενος και ο κύριος ε, Σούριαν. Στις 26 Νοεμβρίου λοιπόν θα γίνει η συνεδρίαση αυτή προκειμένου να ακούσουμε τους ε, θρησκευτικούς αυτούς φιλοσοφικούς και μη ομολογιακούς οργανισμούς. Στόχος είναι να καταφέρουμε να δυναμώσουμε την ευρωπαϊκή δημοκρατία καθώς επίσης και τη συμμετοχή των Ευρωπαίων πολιτών και καταλαβαίνετε ότι η πρωτοβουλία αυτή είναι σημαντική εν ώψη των μελλοντικών ευρωπαϊκών εκλεγών. Πιστεύω ότι μέσω του σεμιναρίου αυτού θα καταφέρουμε να εντείνουμε περισσότερο τη συμμετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι ο πρόεδρος Σούλτς θα έρθει σε επαφή με ορισμένου συντονιστέ προσωρινά, ε, προσωπικά με συγχωρείτε, προκειμένου να συμμετέχουν άμεσα κι αυτοί με παρεμβάσεις στο σεμινάριο αυτό. Επίσης, μια αντιπροσωπεία μας θα πάει στην Ουάσιγκτον από τις 28 στις 31 Οκτωβρίου, προκειμένου να έρθουμε σε επαφή με μέλη του Κογκρέσου, καθώς επίσης και με εκπροσώπους του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, καθώς επίσης και με τις ε, αρχές ε, μιας πολιτείας στις ΗΠΑ. Θα συμμετέχω εγώ στην αντιπροσωπεία αυτή, αλλά και εκ μέρους του ΕΛΚΑ, οι Ταρκόφσκι, Λαμασούρ και Σέφλιν, η Γκουρμά Γκερέρο από τους Σαλιστές, ε, Τερμάκη από το Άλντε, Χέφνερ από τους Πρασίνους και Σόλτς από την Κούε. Θα θυμάστε επίσης ότι η ψηφοφορία για την έκθεση Ταρκόφσκι, η οποία τροποποιεί το άρθρο 81 του κανονισμού, αναβλήθηκε για τις 26 Νοεμβρίου, για τη διάσκεψη των Πρόεδρων των Επιτροπών θεώρησε ότι μέχρι τις 10 Οκτωβρίου οι υπόλοιπες κοινοβουλευτικέ επιτροπές θα μας είχαν διαβιβάσει τις γνωμοδοτήσεις τους. Όντως λάβαμε τις γνωμοδοτήσεις αυτές από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων Διεθνούς Εμπορίου Απασχόλησης και Ανάπτυξης. Δόθηκαν οι γνωμοδοτήσεις αυτές στους συζητητές και στους σκιώδεις συζητητές. Πρέπει όμως να συζητήσουμε αποτελεσματικά και τις γνωμοδοτήσεις αυτές, επομένως αποφάσισα να παρατείνω την προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών μέχρι τις 5 Νοεμβρίου. Όσον αφορά λοιπόν την έκθεση Ταρασκόφσκι, τροποποίηση του άρθρου 81 του κανονισμού, Προβλέπεται λοιπόν συζήτηση για την έκθεση αυτή στην ημερήσια διάταξη της, 26, της 26 Νοεμβρίου και η νέα προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών είναι η 5η Νοεμβρίου. Ξέρετε ότι στο φάκελό σας ο συνήθως έχετε και ένα επικαιροποιημένο ημερωτικό έγγραφο από τις ε, υπηρεσίες μας όσον αφορά τη δικασία επικύρωσης των ε, συνθήκων από τα κράτη-μέλη και αναφέρομαι εδώ πέρα στην έγκριση της ε, συνθήκης για την οικονομική διακυβέρνηση καθώς επίσης και την προσχώρηση της Κροατίας. Μπορείτε λοιπόν να δείτε και το έγγραφο αυτό. Περνάμε τώρα στο σημείο 3 της ημερήσιας διάταξης. που έχει τον εξή τίτλο «Ενιαίοι κανόνες και διαδικασία για την εξυγίανση πιστοτικών ενδρυμάτων και επενδυτικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο ενός ενιαίου μηχανισμού εξυγίανσης και ενός μελλοντικού ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης των Τραπεζών». Έχουμε αναθέσει, όπως ακούσατε, την κυρία Λεγκρή, συντάκτρια γνωμοδότησης για το ζήτημα αυτό και πρέπει να ξεκινήσουμε ευθύ αμέσω τις εργασίες μας, γιατί το χρονοδιάγραμμα της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής μας επιβάλλει να εγκρίνουμε τη δική μας γνωμοδότηση προτού γίνει ψηφοφορία στην Επιτροπή ΕΚΟΝ. Σας προτείνω λοιπόν να δώσουμε στην κυρία Λεγκρίπ ευθύ αμέσω το λόγο. Παρακαλώ. Euh, Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, όντω η Επιτροπή μας έχει αναλάβει τη γνωμοδότηση, την οποία κατόπιν πρέπει να στείλει στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρόκειται για το θέμα της Τραπεζικής Ένωσης, το δεύτερο πυλώνα της Τραπεζικής Ένωσης πιο συγκεκριμένα. Η δημιουργία της Τραπεζικής Ένωσης αποτελεί τμήμα της ενίσχυσης της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, κατά την άποψή μου μια απαραίτητη βαθμίδα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Έχουμε ξεκινήσει τις εργασίες μας για μία σειρά μέτρων με σκοπό την σταθεροποίηση και την ενίσχυση της ε, δεοντολογίας, την επιστροφή της εμπιστοσύνης των ε, πολιτών, των αγορών, ε, κάτι πολύ δύσκολο, και να ε, βελτιωθεί το κλίμα το οποίο έχει επιδεινωθεί κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Προσπαθούμε επίσης να οδηγήσουμε στην ανάκαμψη έτσι ώστε οι υπηρεσίες της ε, εσωτερικής αγοράς, οι υπηρεσίες στον τομέα των τραπεζικών να εξηγιανθούν. Υπάρχει σήμερα μία ανησυχία, μία έλλειψη εμπιστοσύνης από το ένα εθνικό σύστημα στο άλλο. Υπάρχει ο φόβος ε, ότι τα προβλήματα μπορεί να επεκταθούν. Γι' αυτό και σήμερα προσπαθούμε να δημιουργήσουμε κοινού κανόνες και μια ε, ευρωπαϊκή ταυτότητα για τις τράπεζες που είναι παρούσες σε πάνω από μια ευρωπαϊκή χώρα. Ασχολούμαστε λοιπόν ιδιαίτερα σε αυτή τη γνωμοδότηση με τις τραπεζικές υπηρεσίες με σκοπό μελλοντικά προβλήματα στα τραπεζικά συστήματα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με ενιαίο τρόπο και με μια ενιαία, ελπίζουμε, λήψη αποφάσεων η οποία θα βελτιώσει την αντίδραση και θα την κάνει ταχύτερη. Αναφέρομαι λοιπόν πολύ συγκεκριμένα σε αυτό το δεύτερο πυλώνα της ε, Τραπεζικής Ένωσης, μια πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εμείς η Επιτροπή μας ε, καλείται να γνωμοδοτήσει, είμαι η συγκίτρια για τη γνωμοδότηση αυτή, με σκοπό να επεξεργαστούμε το θεσμικό πλαίσιο εντός του οποίου καλείται να λειτουργήσει αυτή η Τραπεζική Ένωση και τα διάφορα όργανα καθώς και ο μηχανισμός και το ταμείο. Αυτός λοιπόν ο ενιαίος μηχανισμός εξυγίανσης και ε, το Ταμείο έχει σαν σκοπό να αντιμετωπίσει μελλοντικές κρίσεις με έναν ολοκληρωμένο μηχανισμό εξυγίανσης. Με σκοπό να δημιουργηθεί ένα Συμβούλιο Εξυγένσης με τη συμμετοχή των κρατών μελών βεβαίως και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτός ο νέος μηχανισμός βεβαίως δημιουργεί ερωτηματικά θεσμικού χαρακτήρα. Η δική μας Επιτροπή στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της καλείται να απαντήσει σε αυτές τις ε, ερωτήσεις καθώς και σε όλα τα ε, θέματα που απορρέουν όπως παραδείγματο χάρη αυτό του δημοκρατικού ελέγχου. Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι η νομική βάση επί της οποίας στηρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το άρθρο 114 της Συνθήκης το άρθρο 114 που προβλέπει την υιοθέτηση μέτρων που έχουν σχέση την ενοποίηση των εθνικών διατάξεων για τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Εγώ θεωρώ ότι αυτή η νομική βάση είναι ορθή και μπορεί να αντιμετωπίσει τελικά τον τελικό στόχο που είναι η διακυβέρνηση, ο μηχανισμός και ε, το ταμείο το οποίο θα πρέπει να βρίσκεται στο εσωτερικό του θεσμικού πλαισίου, όπως προβλέπεται από τις συνθήκες. Αυτή λοιπόν η νομική βάση για αυτόν τον κανονισμό θα πρέπει να λάβει υπόψη του και το σημείο 6 του ψηφίσματος που πέρασε από την Ολομέλεια τον Σεπτέμβριο του 2012 και αφορά την Τραπεζική Ένωση. Αυτό το σημείο 6 λοιπόν αναφέρει ότι κάθε αλλαγή στην εποπτεία, καθώς και η μεταφορά αρμοδιοτήτων σε άλλα θεσμικά όργανα, θα πρέπει να ε, ακολουθείται από αντίστοιχη πρόοδο στην διαφάνεια και σε αντίστοιχα δικαιώματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα πρέπει να μπορεί να θέσει ερωτήσεις και να αμφισβητήσει κάποιες αποφάσεις. Σε ένα ψήφισμα λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Ολομέλεια το Σεπτέμβριο του 2012 αναφέρθηκε σε αυτό ακριβώς το σημείο. Εγώ βασίστηκα σε αυτό στην εργασία μου. Περισσότερη διαφάνεια λοιπόν, περισσότερες αρμοδιότητες για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έτσι ώστε να μπορέσει να ασκηθεί δημοκρατικός ε, κοινοβουλευτικός έλεγχος. Σας προτείνω λοιπόν κάποιες τροπολογίες οι οποίες επικεντρώνονται σε τρία σημεία με σκοπό τη βελτίωση της αρχικής πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αρχικά λοιπόν σας ζητώ να ξαναδούμε το τρίτο τμήμα που αφορά το θεσμικό πλαίσιο κάνοντας ε, μια συγχώνευση του τίτλου 1 και 4 για καλύτερη αν θέλετε συνοχή στην παρουσίαση των προτάσεων. Μου φάνηκε λοιπόν απαραίτητο να ενισχύσουμε τον κοινοβουλευτικό έλεγχο όσον αφορά τις αρμοδιότητες εξυγίανσης αυτού του Συμβουλίου. Τρίτο σημείο που με απασχόλησε και σε αυτό αναφέρονται και διάφορες άλλες τροπολογίες είναι η ενίσχυση του δημοκρατικού χαρακτήρα αυτής της νέας υπηρεσίας που θα πρέπει να συμμετέχουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλιο. Ενίσχυση λοιπόν του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τις δυνατότητες εξυγίανσης, αυτού του Συμβουλίου Εξυγίανσης, που πρέπει να υπάρξει λοιπόν έγκριση, επαναλαμβάνω έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις αποφάσεις αυτού του Συμβουλίου. Τροπολογίες 4, 37 και 40. Ζητώ επίσης ενίσχυση του κοινοβουλευτικού ελέγχου με ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αυτού του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή μεταξύ των Προέδρων και Αντιπροέδρων ε, των Αρμόδιων Επιτροπών. Τροπολογία 16 και 18. Η άλλη όψη του νομίσματος αυτού του κοινοβουλευτικού δημοκρατικού ελέγχου είναι, ανάλογα βεβαίως με το πρωτόκολλο 1 που προσαρτημένο και εδώ αναφέρομαι στα άρθρα 69, 70, 71 και 352 της συνθήκης για την συμμετοχή των θεσμικών οργάνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, σε αυτήν την προσπάθεια εξυγένσης. Ζητώ λοιπόν το Συμβούλιο εξυγίανσης να στέλνει το πρόγραμμα εργασιών του στο Κοινοβούλιο, τροπολογία 22 επίσης, τα θεσμικά όργανα και το Κοινοβούλιο να μπορούν να στέλνουν ε, παρατηρήσεις ε, στο Συμβούλιο, τροπολογία 15, τροπολογία τώρα 41 και 42, το Συμβούλιο να στέλνει τους ε, λογαριασμούς του ετήσιους λογαριασμού του για το οικονομικό έτος που θα ακολουθήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η γνωμοδότηση λοιπόν θα πρέπει να περιορίζεται και να στοχεύει τις αρμοδιότητες της δικής μας ε, Επιτροπής. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει εδώ να ασχοληθούμε με όλα, όλες τις πτυχές της Τραπεζικής Ένωσης και του δεύτερου πυλώνα της αλλά όσον αφορά τις δικές μας αρμοδιότητες και την ενίσχυση του δημοκρατικού ελέγχου και την άσκηση του δημοκρατικού ελέγχου σας υποβάλλω αυτή τη γνωμοδότηση. Δεν θα σας παρουσιάσω με περισσότερες λεπτομέρειες της τροπολογίας, αλλά είμαι στη διάθεσή σας για να συζητήσουμε τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά σας έτσι ώστε να επεξεργαστούμε περαιτέρω αυτή την γνωμοδότηση, να την ολοκληρώσουμε. Νομίζω ότι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών δεν έχει ακόμα καθοριστεί, αλλά σκοπός μας είναι να είναι σύντομη αυτή η προθεσμία έτσι ώστε να μπορέσουμε να ψηφίσουμε στις 25 Νοεμβρίου, Δευτέρα 25 Νοεμβρίου. Δηλαδή την προηγουμένη της ημέρας που θα ψηφίσει η Οικονομική Επιτροπή. Σας ευχαριστώ πολύ και βεβαίως με χαρά θα ακούσω τις παρατηρήσεις σας. Σας ευχαριστούμε κυρία Λεγκρίπ για την γνωμοδότησή σας, για την παρουσίαση αυτή και για την τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάσατε και συντάξατε την γνωμοδότηση αυτή τόσο γρήγορα, ενώ δεν είχατε πάρα πολύ χρόνο στην διάθεσή σας. Μπορούμε να ξεκινήσουμε τώρα τη συζήτηση για την γνωμοδότηση αυτή. Δεν ξέρω αν θέλει να πάρει κάποιο το λόγο. Κύριο κύριος Νταφ. Um, yes. Ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Πρέπει πραγματικά να χειριστούμε μεγάλη προσοχή για αυτό το ζήτημα. Γιατί είναι μια κίνηση άνευ από πλευράς των ευρωπαϊκών οργάνων για την εποπτεία του τραπεζικού συστήματος Ευρωπαϊκής Ένωσης με σημαντικές συνέπειες για τι ανεξαρτησία, αν θέλετε, και την ε, αυτοκυριαρχία των κρατών μελών και την ακαιρεότητα των τραπεζών. Θα ήθελα να ρωτήσω αν έχουμε λάβει ήδη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για αυτό το θέμα. Γιατί εάν δεν την έχουμε λάβει, θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι να την ε, λάβουμε. Δεύτερον, παρακολουθώ με προσοχή παρακολούθησα με προσοχή την, προσοχή, την ε, παρουσίαση της κυρίας Ελεγκρίπ, την οποία και ευχαριστώ. Βλέπω όμως ότι προσπαθεί να προαγάγει το ρόλο των Ευρωπαϊκών Εθνικών Κοινοβουλίων για αυτό το ζήτημα και για να είμαι το σαφή, θα πρέπει να μελετήσουμε αναλυτικά τις ε, τροπολογίες που μας προτείνει. για να δούμε ότι υπάρχει σωστή ενημέρωση προς τα εθνικά κοινοβούλια για τη διαχείριση αυτού του νέου ε, εποπτικού συστήματος. Όμως, εφόσον μιλάμε για ενιαίο εποπτικό μηχανισμό και με ενιαίο μηχανισμό εξυγίανσης, είναι σημαντικό τα εθνικά κοινοβούλια να μην συμμετέχουν στην νομοθετική διαδικασία. Το προσχέδιο λοιπόν χρήζει προσεκτικής μελέτης πριν καταφέρει τουλάχιστον πιστή τουλάχιστον η Επιτροπή Λίβε ότι βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο. Και πρέπει να δούμε και την αντίστοιχη προθεσμία των Μητροπολιγιών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Ντάφα. Ξέρετε ότι η εισηγήτρια ήδη μίλησε για την προθεσμία αυτή, με πρόλαβε ουσιαστικά. Ξέρετε ότι πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα γιατί η Επιτροπή ΕΚΟΝ πρέπει και αυτή οριστικά στις 26 Νοεμβρίου να εγκρίνει την έκθεσή της. Άρα εμείς μέχρι τις 25 θα πρέπει να έχουμε εγκρίνει την γνωμοδότησή μας. Άρα, όντω μπορούμε να πούμε ότι η ημερομηνία κατάθεση τροπολογιών, η προθεσμία δηλαδή, θα είναι η 5η Νοεμβρίου. Δεν έχουμε λοιπόν πολύ χρόνο στη διάθεσή μα και όντω ο κύριο Ντάφ έχει απόλυτο δίκιο στα όσα λέει. Πρέπει λοιπόν να εργαστούμε πάρα πολύ σκληρά, πάρα πολύ έντονα, προκειμένου να καταφέρουμε να εγκρίνουμε και εμεί την γνωμότηση αυτή πολύ σύντομα. Κύριο Γκουαλτιέρη έχει το λόγο. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ξέρετε ότι θα έχουμε τη δυνατότητα με την εισηγήτρια και εμεί οι σκιώδη εισηγητέ ε, να παρουσιάσουμε καλύτερα και με περισσότερε λεπτομέρειε ε, τι δικέ μα τι θέσει. Ξέρετε ότι ε, λάβαμε πριν από λίγο ουσιαστικά το σχέδιο γνωμοδότησης της κυρίας Λεγκρίπ. Ξέρετε ότι το ζήτημα είναι πάρα πολύ πολύπλοκο και επομένως πρέπει να αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο για να μελετήσουμε το έγγραφο αυτό. Θα περιοριστώ σε κάποιες σύντομες παρατηρήσεις προκαταρκτικές σε σχέση με τα όσα είπε η κυρία Λεγκρίπ. Καταρχάς, εκτιμώ ιδιαίτερα προφανώς την ταχύτητα με την οποία εργάστηκε η κυρία Λεγκρίπ. Θαυμάζω ουσιαστικά την ταχύτητα αυτή με την οποία εργάστηκε, αλλά θα ήθελα πραγματικά να υποστηρίξω και ουσιαστικά τη δική της τη θέση, ότι δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει μια νομική βάση για τον κανονισμό αυτό. Το ζήτημα είναι αρκετά αμφιλεγόμενο και μολονότι από τεχνικής πλευράς Μπορούμε να πούμε ότι είναι δύσκολο να καταφέρουμε μέσω τροπολογιών να αναδείξουμε το ζήτημα αυτό, πάντως είναι πάρα πολύ σημαντικό η δική μας Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων να εκφραστεί με απόλυτη σαφήνεια για το ζήτημα αυτό, της νομικής δηλαδή βάσης. Και όπως είπε η κυρία Λεγκρίπα, είναι σημαντικό να εγκρίνουμε ως νομική βάση το άρθρο 114 της Συνθήκης, ιδίως υπό το φως του ουσιαστικότατου ουσιαστικότατου θεμελιώδους ρόλου που θα διαδραματίζει ένας τέτοιος ενιαίος μηχανισμός εξυγίανσης όσον αφορά μια αποτελεσματική, αποδοτική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Εκ πρώτης όψεως, νομίζω ότι είναι πολύ θετικές οι τροπολογίες εκείνες που έχουν ως στόχο να αυξήσουν το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ξέρετε ότι υπάρχει και ένα πολύ σημαντικό προηγούμενο όσον αφορά δηλαδή την διαδικασία διαβούλευσης που είχαμε στο παρελθόν, όπου απλώς συμμετείχε σε διαβούλευση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ξέρετε ότι καταφέραμε ως Κοινοβούλιο να αυξήσουμε, να δυναμώσουμε το ρόλο μας στα πλαίσια της λειτουργίας του ενιαίου μηχανισμού εποπτείας και συνεπώς Εφόσον βρισκόμαστε πλέον στη συνήθινη νομοθετική διαδικασία, δηλαδή στη συναπόφαση, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ενισχύεται ο ρόλος και συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρέπει επίσης να σας πω ότι θα υπάρχουν και πολύ σημαντικές επιπτώσεις από τον ενισχυμένο αυτό ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον ενιαίο μηχανισμό εξυγίανση, καθώ επίση και στον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό και θα υπάρχουν συνέχεια επιπτώσει και στην λεγόμενη πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να νομιμοποιείται πλήρω να συμμετέχει στη νέα αυτή οικονομική διακυβέρνηση κάθε φορά που προβλέπονται νέα μέτρα τα οποία εμπλέκουν εν μέρη τα κράτη-μέλη. Όσον αφορά λοιπόν το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη νέα πολυεπίπεδη οικονομική κυβέρνηση, είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι από τη μια πλευρά έχουμε εδώ πέρα μία διαδικασία όπου βλέπουμε ότι η Ευρωζώνη ανοίγεται περισσότερο και θελός προς τα κράτη-μέλη, όσοι επιθυμούν δηλαδή να εισχωρήσουν σε αυτήν, και από την άλλη όμως προβλέπεται και ένα συγκεκριμένο σύστημα ελέγχου τον οποίο έλεγχο θα διδραματίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μολονότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια δυσανάλογη συμμετοχή των κρατών μελών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στους ενίους μηχανισμούς, τόσο τον μηχανισμό εξυγίανσης όσο και τον μηχανισμό εποπτείας. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμμετέχει ενεργά στα δύο αυτά συστήματα, χωρίς να προβλέπεται αναγκαστικά η συμμετοχή επιπλέον ξένων φορέων. Είναι πολύ σημαντικές λοιπόν οι παρατηρήσεις που κάνει η κυρία Λεγκρίπη για το ζήτημα αυτό, αλλά πολύ θετικέ είναι επίσης και οι παρατηρήσεις της όσον αφορά την ε, πολιτική που θα ακολουθήσει γενικότερη Ευρωπαϊκή Ένωση για τους ε, μηχανισμούς οικονομικής εποπτείας. Τώρα, η διπλή αυτή νομιμοποίηση της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά δηλαδή τους πολίτες και όσον αφορά τα κράτη-μέλη και όσον αφορά ουσιαστικά τα δύο όργανα εκπροσώπησης, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο. Είπαμε ότι ως προς αυτό θα πρέπει να αυξήσουμε το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και γι' αυτό το λόγο επιφυλάσσουμε και εγώ όπως και ο συνάδελφος Νταφ να εξετάσουμε καλύτερα τις προτάσεις της κυρίας Λεγκρίπ. Σε μια πρώτη φάση θα έλεγα ότι θα πρέπει να είμαστε κάπως προσεκτικοί όσον αφορά την άμεση συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων στον ενιαίο μηχανισμό εξυγίανσης. Είμαι κάπως διστακτικός απέναντι σε αυτό. Δεν λέω ότι δεν μπορούν τα εθνικά κοινοβούλια να έχουν και αυτά ένα ρόλο όσον αφορά την ευρωπαϊκή νομοθετική διαδικασία, όπως άλλωστε προβλέπεται από τη συνθήκη και τα σχετικά πρωτόκολλα. Αυτό το οποίο λέω είναι ότι ε, τα εθνικά αυτά κοινοβούλια έχουν βέβαια ως ε, ρόλο να ελέγχουν τις εθνικές κυβερνήσεις. Πρέπει επίσης να δημιουργούν διάβλους διαλόγου μεταξύ των πολιτών και των κυβερνήσεων, αλλά το να συμμετέχουν επιπλέον και σε νέους μηχανισμούς όπως ο μηχανισμός εξυγίανσης και ο εποπτικός μηχανισμός ενδεχομένως να είναι κάπως υπερβολικό και τελικά να περιπλέκει κάπως περαιτέρω και τον ρόλο που έχουν τα εθνικά κοινοβούλια. Νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να κάνουμε μία μνήα στα εθνικά κοινοβούλια χωρίς να επιμένουμε τόσο πολύ όσο κυρία Λεγκρίπ. Τέλος, ένα ερώτημα που θέλω να θέσω προς τη συνάδελφο Λεγκρίπ. Νομίζω ότι ε, λείπουν κάποιες τροπολογίες όσον αφορά τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου αυτού. Αυτό τι σημαίνει, ότι ενδεχομένως να έχουμε μία επικριτική στάση απέναντι στην στάση μας υπηρεσία υπηρεσία για την υπόθεση Μερώνη όσον αφορά το ρόλο που θα μπορούσε να έχει το Συμβούλιο αυτό. Επομένως θεωρεί η κυρία Λεγκρίπ ότι τα όσα μας είπε η νομική υπηρεσία του Συμβουλίου δεν είναι τελικά δικαιολογημένα, μήπως είναι κάπως υπερβολικά και ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αντίθεση με το Συμβούλιο δεν θα πρέπει να δίνει αρμοδιότητες διακριτικής ευχέρειας πιο υπερβολικές από αυτές που προβλέπονται από το θεσμικό όργανο που υποβάλλει τις αρμοδιότητες αυτές, που εκχωρεί τις αρμοδιότητες αυτές. Και το ζήτημα αυτό είναι ιδιαίτερα λεπτό και νομίζω ότι θα πρέπει να επανέλθουμε στο ζήτημα αυτό. Νομίζω ότι η δική μας Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει τροπολογίες, να αποφανθεί για το ζήτημα αυτό, το ρόλο δηλαδή της αρμοδιότητας του Συμβουλίου, όπως επίσης πρέπει να το κάνει και για το ζήτημα της νομικής βάσης και νομίζω ότι κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε τελικά να επηρεάσουμε την όλη πορεία που θα ακολουθήσει ο κανονισμός αυτός. Ο κύριος Μπρόνς έχει τώρα το λόγο. Ε, Ευχαριστώ. Εκ πρώτης όψεως θα μπορούσε κανείς να νομίζει ότι έχει οικονομικούς στόχους η πρόταση. Και το οργανικό οικοδόμημα, το θεσμικό οικοδόμημα είναι μόνο ένα σύνολο ε, πολιτικών ε, δομών που επιτυχάνουν αυτούς τους στόχους. Όμως, αν εξετάσουμε πιο προσεκτικά ακούγοντα και τις ξεκάθαρες εξηγήσεις ε, της εισηγήτριας, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ίσως να ισχύει και το αντίθετο. Στη δεύτερη τρίτη παράγραφο αναφέρεται ότι είναι πολύ σημαντικό να ε, αυτή η σύνδεση μεταξύ ε, τραπεζών και κρατών. Και σήμερα μάλιστα είπαμε ότι είναι πολύ σημαντική η Τραπεζική Ένωση για την, ολοκλήρωση, για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, αλλά και η βελτίωση της λειτουργία ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει πολύ σημαντικό ρόλο. Πράγματι, η συγγήτρια ανέφερε το ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων, όμως ε, βάσει της υποδοχής που ακούσαμε σήμερα, φαίνεται ότι αυτό δεν πρέπει να συμβεί. Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι ο βασικός ε, στόχος και οποιοδήποτε οικονομικό προτέρημα ε, είναι εντελώ τυχαίο. Αλλά εντάξει, δεν θέλω να επεκταθώ. Σίγουρα θα υπάρχουν και κάποιοι πολίτες που μας παρακολουθούν, ε, όμως ε, μπορεί εκείνοι να διαφωνήσουν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε, κύριο Σέφνερ. Äh, Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν να ευχαριστήσω την κυρία Ντεγκρίπ, γιατί είναι πάρα πολύ χρήσιμη και απαραίτητη αυτή η πρόταση που μας παρουσίασε σήμερα. Όντως μας πιέζει ο χρόνος και πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει να εργαστούμε γρήγορα Συμφωνώ όμως και με το συνάδελφο Νταφ και τον κύριο Γκαλτιέρη. Υπάρχουν κάποια θέματα νομικά, υπάρχουν κάποια θέματα που ενδεχομένως θα πρέπει να τα επεξεργαστούμε γιατί έχουν συνέπειες και πολιτικές έχουν συζητηθεί από ακαδημαϊκούς, από πολιτικούς, σε αρκετά κράτη-μέλη έχει προκαλέσει συζήτηση το θέμα αυτό. Δεν μπορούμε λοιπόν τόσο εύκολα να το αντιμετωπίσουμε το θέμα της νομικής βάσης, το θέμα του δημοκρατικού ελέγχου, το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κατά την άποψή μου θα πρέπει ίσως να το προσέξουμε λίγο περισσότερο. Και αυτό που είναι σημαντικό για μας είναι να μας δοθεί το κείμενο όχι μόνο στα γαλλικά. Με την έννοια ότι για να το συζητήσουμε και να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε όλες αυτές τις πτυχές τις οποίες σας ανέφερα, χρήσιμο θα ήταν και να το έχουμε στη γλώσσα μας το κείμενο, αλλά και να περιμένουμε και την νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου την τοποθέτησή της. Για μένα η γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας του Κοινοβουλίου είναι απαραίτητη και θα μας διευκολύνει πάρα πολύ την εργασία μας. Αυτά. Δεν ξέρω τι κατεύθυνση θα πάρει αυτή η συζήτηση, αλλά προηγουμένως θα πρέπει είναι προϋπόθεση για μένα να έχουμε το κείμενο σε όλες τις γλώσσες για να μπορέσουμε να το συζητήσουμε. Να δώσω στην κυρία Λεγκρίπ τώρα το λόγο για να απαντήσει. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ για τις παρεμβάσεις σας και έχετε δίκιο όταν λέτε ότι η ταχύτητα με την οποία επεξεργάστηκα αυτό το σχέδιο, γιατί προς το παρόν ε, πρόκειται για σχέδιο γνωμοδότησης, σίγουρα αυτό προκάλεσε κάποιες αδυναμίες, κάποιες ελλείψεις. Για άλλη μια φορά ο χρόνος μας πιέζει και γνωρίζω ότι χρειάζεται περισσότερη επεξεργασία σε όλες τις πτυχές εξαλλού του θέματος αυτού. Άκουσα πολύ προσεκτικά και τον κύριο Νταφ, Καλτιέρη και Χέφνερ όσον αφορά τις αρμοδιότητες για τα Εθνικά Κοινοβούλια. Εγώ σε καμία περίπτωση δεν ήθελα να προτείνω κάποια παρέμβαση στις νομοθετικές διαδικασίες, αλλά αναφερόμουν μάλλον σε ανταλλαγή πληροφοριών. Σίγουρα λοιπόν εδώ άκουσα αυτό που είπατε και πρέπει να επεξεργαστούμε περαιτέρω το κείμενο και να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στην διατύπωσή μας. Ακριβώς γιατί αυτό το θέμα σίγουρα είναι αρκετά ευαίσθητο. Κύριε Πρόεδρε, εγώ σαφώς και είμαι υπέρ του να ζητήσουμε γνωμοδότηση από την νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου. Ιδιαίτερα αν αυτό το ζητούν ε, κάποιες πολιτικές ομάδες. Εγώ συμφωνώ με αυτήν την πρόταση, ε, λαμβάνοντας βεβαίω υπόψη την πάρα πολύ σύντομη διαδικασία την οποία μας έχετε προτείνει, αλλά βεβαίως μια τέτοια συμβολή της νομικής υπηρεσίας θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμη. Αυτά προς το παρόν τουλάχιστον και βεβαίως με μεγάλη χαρά θα συνεχίσω την ε, επεξεργασία αυτού του σχεδίου γνωμοδότησης μαζί σας με την απαραίτητη βεβαίω ταχύτητα. Σας ευχαριστούμε κυρία Λεγκρίπ. Θέλει κάποιος στο λόγο, κύριος Νταφ. Euh, euh. Ένα σύντομο ερώτημα προς την εισηγήτρια. Est-ce euh, περιμένουμε γνωμοδότηση της Κεντρικής Τράπεζας ή όχι. Κατανοώ ότι το να έχουμε και τη γνωμοδότηση της Κεντρικής Τράπεζας θα ήταν πραγματικά πολύ σημαντικό. Όμως, για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω καμία ιδέα ε, πότε θα μπορούσε να μας αποσταλεί τέτοια γνωμοδότηση. Δεν έχει προσδιοριστεί κάτι τέτοιο. Τώρα, αν αυτό θα μας ε, εμποδίσει ε, στο ρυθμό ε, των εργασιών μας πολύ ή λιγότερο, νομίζω ότι εμείς θα πρέπει να προχωρήσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα και βεβαίως αν αυτό γίνει σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα θα ήταν πολύ θετικό το να έχουμε και την γνωμοδότηση της ΕΚΤ. E Μάλιστα, κι άλλοι θέλουν τώρα την, το λόγο, ο κύριος Γκουαλτιέρη. Κύριε Πρόεδρε, μία σύντομη παρατήρηση όσον αφορά τα ο κύριο Ντάφα μόλις πριν από λίγο. Και εγώ νομίζω θα ήταν πολύ ενδιαφέρον και πολύ σημαντικό να διαθέτουμε τη γνωμοδότηση Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αλλά ξέρετε, ακολουθούμε τη συνήθη νομοθετική διαδικασία. Είμαστε δηλαδή συνομοθέτες. Έτσι λοιπόν, αν η γνωμοδότηση αυτή φτάσει εγκαίρως, τόσο το καλύτερο. Ωστόσο, νομίζω ότι δεν πρέπει εμείς να περιμένουμε την γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για να προχωρήσουμε με το νομοθετικό μας έργο. Ξέρετε ότι θα πρέπει και εμείς να ολοκληρώσουμε την εξέταση του κανονισμού αυτού εγκαίρως, δηλαδή πριν λάβουν χώρα οι επόμενες ευρωπαϊκές εκλογές. Δηλαδή θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι σε πρώτη ανάγνωση, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι η γνωμοδότηση της Επιτροπής μας θα πρέπει εγκαίρως να εγκριθεί, προκειμένου να εγκριθεί και η έκθεση της καθήλυνα αρμόδιας Επιτροπής, θα ακολουθήσει τριμερής διάλογος και ούτω Θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να εμπλέξουμε νέα στοιχεία αυτή τη στιγμή στη διαδικασία που θα περιπλέξουν περισσότερο τα πράγματα. Αν μπορούμε να έχουμε γρήγορα τη γνωμοδότηση τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αυτό θα ήταν θετικό. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει η γνωμοδότηση τη ΕΚΤ να γίνει προπόθεση για να συνεχίσουμε εμεί το έργο μα για αυτή την έκθεση. Allora, ε, mi pare... Πρόεδρος, νομίζω ότι μπορούμε να ολοκληρώσουμε το σημείο αυτό. Από τη συζήτηση φάνηκε ότι όντω το ζήτημα είναι ιδιαίτερα λεπτό. Μας απασχολεί το ζήτημα της νομικής βάσης, το ζήτημα της αρμοδιότητας των εθνικών κοινοβουλίων, το ζήτημα της ε, αρμοδιότητας των αρμοδιοτήτων του board. Νομίζω λοιπόν ότι ε, τα ζητήματα αυτά θα πρέπει να έχουν την πλήρη προσοχή μας και θα πρέπει να εμβανθύνουμε όσο δυνατόν περισσότερο. Μας πιέζει όμως και ο χρόνος και ξέρετε ότι α, τον τελικό λόγο θα έχει η Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων. Την επόμενη Πέμπτη θα έχουμε μια συνάντηση με την πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικών, την κυρία Μπόλς, η οποία ζήτησε να υποβάλει μια γνωμοδότηση όσον αφορά την έκθεση Ταρκόφσκι για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Θα μπορούσαμε λοιπόν στην συνάντηση αυτή να τη ζητήσουμε λίγο περισσότερο χρόνο. Και αυτό γιατί η γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όπως και γενικότερα όλες οι γνωμοδοτήσεις από τις νομικές υπηρεσίες, αλλά αυτή συγκεκριμένη από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δεν ενδιαφέρει μόνο εμάς, αλλά ενδιαφέρει κυρίως, θα έλεγα, την Επιτροπή Νομισματικής και Οικονομικής Πολιτικής. Ενδεχομένως λοιπόν και η ίδια η Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής να αποφασίσει τελικά να δώσει περισσότερο χρόνο στην εξέταση αυτής της έκθεσης προκειμένου να παραλάβει και αυτή τη γνωμοδότηση της ΕΚΤ. Πάντως μέχρι στιγμής προβλέπεται η έγκριση της σχετικής έκθεσης από την ΕΚΟΝ στις 26 Νοεμβρίου, εμείς θα πρέπει να έχουμε ολοκληρώσει την ψηφοφορία μας μέχρι τις 25 Νοεμβρίου. Προθεσμία κατάθεσης λοιπόν τροπολογιών η 5η Νοεμβρίου. Είναι όμως προσωρινές όλες αυτές οι ημερομηνίε και μπορεί ενδεχομένως να δώσουμε μια παράταση. Εφόσον βέβαια μας το επιτρέψει αυτό η Επιτροπή ΕΚΟΝ. Περιμένουμε τώρα και να ξεκινήσουμε και τις ψηφοφορίες ή μάλλον ο κύριος Σέφνερ θέλει το λόγο. Παρακαλώ. Ε, όταν ζήτησα αυτή τη γνωμοδότηση της ε, νομικής ε, υπηρεσίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό νομίζω ότι μπορούμε να ελέγξουμε τις ε, ημερομηνίες. Αλλά όσον αφορά τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, νομίζω ότι αυτό βεβαίως δεν το ελέγχουμε, αλλά τουλάχιστον κάποιες ενδείξεις θα ήταν χρήσιμες όσον αφορά το πότε θα μας ταλεί richiesta μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό πάλι με την κυρία Μπόλς, την ε, Πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, όταν θα τη συναντήσουμε την επόμενη Πέμπτη. Έχουμε λίγα λεπτά στη διάθεσή μας πρωτού ξεκινήσουμε της ε, ψηφοφορίας και θα ζητήσω λοιπόν από τον συνάδελφο Μέσερμιτ, ο οποίος κάθεται εδώ πέρα, στα δεξιά μου και το τον είχα δει, αν θα μπορούσε να μας μιλήσει πολύ σύντομα για το ζήτημα του προπολογισμού, καθότι είναι αρμόδιος για το ζήτημα αυτό. Thank you, Chair. Yes, I... Uh, Ευχαριστώ. Όπως ξέρετε, ψηφίσαμε ομόφωνα υπέρ μια, του, της νομοδότησης για τον προπολογισμό από την ΑΦΚΟ. Δεν έχει γίνει ακόμα ψηφοφορία στην Επιτροπή Προπολογισμού. Τα μέλη όμως έχουν υιοθετήσει όλες τις ε, τροπολογίες εκτός ε, δύο. Και αυτές οι δύο που δεν υιοθετήθηκαν ήταν η 69.00 ε, για την προσθήκη δύο παραγράφων για τις επερχόμενε ευρωπαϊκές εκλογές του χρόνου και δεύτερον 6903 για νέα γραμμή προπολογισμού για την εφαρμογή της ε, πρωτοβουλία για τους πολίτες. Από είχαμε πολλά τεχνικά προβλήματα και θέματα με την πρωτοβουλία αυτή και ζητήσαμε να ψηφιστούν για τον επόμενο προπολογισμό. Αυτές οι δύο τροπολογίες λοιπόν από την Επιτροπή μου δεν εγκρίθηκαν για τον προπολογισμό. Ενημέρωσα τη γραμματεία ότι θα πρέπει αυτές οι δύο ανεξάρτητες τροπολογίες να παρουσιαστούν στην ψηφοφορία στην Ολομέλεια και ελπίζω και εσείς ε, να τη στηρίξετε. Αυτά προς πληροφορήσεις. Σας ευχαριστώ. Ε, Σας ευχαριστούμε κύριε Μέσσερ Σμίτ. Νομίζω τώρα ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε τις πληροφορίες μας. Η πρώτη έκθεση είναι ο Οργανισμό Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Συνεργασία και την Κατάρτιση. Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε. Μπορούμε να έχουμε δύο λεπτά στη διαθεσή μα για να προετοιμαστούμε λίγο για την ψηφοφορία. Ούτω ή άλλω ξεκινάμε λίγο νωρίτερα, έτσι δεν είναι. Πρόεδρο, ναι, προφανώ μπορεί να το ζητήσετε, δεν ξέρω αν θα σα το επιτρέψω, σα το επιτρέπω. Δύο λεπτά. Δύο λεπτά πρωτού ξεκινήσουμε την ψηφοφορία για την Ευρωπόλα. Ναι, ναι, δύο λεπτά πρωτού ξεκινήσει η γενικότερη διαδικασία της ψηφοφορίας. Αυτό σας ζητάω. Για να καταφέρουμε λίγο να οργανωθούμε. Εφόσον τους άλλους λίγο νωρίτερα τις ξεκινάμε τις ψηφοφορίες από ό,τι προβλεπόταν. No, la mia richiesta era di avere una sospensione di Διάλειμμα δύο λεπτών απλώς σας ζήτησα προκειμένου να καταφέρουν όλες οι πολιτικές ομάδες να προετοιμαστούν σε σχέση με τους καταλόγους ψηφοφορίας. Εφόσον τους άλλως ξεκινάμε αυτή τη στιγμή νωρίτερα, δεν έχουμε καθυστέρηση. Ένα λεπτό μόνο δώστε μας για να προετοιμάσουμε τους καταλόγους ψηφοφορίας. Μα δεν ξεκινάμε πλέον νωρίτερα. Έχετε πάντως δύο λεπτά στη διάθεσή σας. Δύο λεπτά διάλειμμα προτού ξεκινήσουμε με τις ψηφοφορίες. Πέρασαν τα δύο λεπτά. Ξεκινάμε με τις ψηφοφορίες. Να σας πω καταρχάς ότι αν εκ πρώτη όψεως δεν είναι σαφής ο αριθμός πλειοψηφίας μειοψηφίας, θα προχωρήσουμε στην ηλεκτρονική επαλήθευση αμέσως και θα γίνει ηλεκτρονική επαλήθευση πάντα για την τελική ψηφοφορία γιατί ε, νομίζω ότι η κατάσταση δεν είναι απαραίτητα ξεκάθαρη για όλες τις εκθέσεις. Θα προχωρήσουμε λοιπόν και θα λειτουργήσουμε αυτόν τον τρόπο. Ας έχετε λοιπόν έτοιμες τις κάρτες σας για τελική ψηφοφορία. Ξεκινάμε με την έκθεση ΤΕΙΝ για την πρόταση κανονισμού όσον αφορά τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία και την Κατάρτιση στον τομέα της επιβολής του νόμου Ευρωπόλου και σχετικά με την τροποποίηση των αποφάσεων 371 του 2009 και 681 του 2005. κυρία Τέιν δεν είναι εδώ. Έχει ενεργημένε υποχρεώσει στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Κύριε Ντάφ, θέλετε το λόγο. Όλα Μπορούμε να ψηφίσουμε ή θέλετε το λόγο. Παρακαλώ. Just one quick... Πολύ σύντομα. για την αιτιολογική σκέψη 6 στο, στη συμβαστική λύση που έχει βρεθεί. Ζητούμε η αναφορά στη ΣΥΠΟΛ να μεταφερθεί και να τεθεί δίπλα στη Europol. Μετά τη σύνταξη και τη διατύπωση, είδαμε ότι η Κορεπέρα αποφάσισε να προτείνει μεταφορά της ΣΥΠΟΛ στην Βουδαπέστη, που από όσο ξέρω εγώ, τις δικές μου γεωγραφικές γνώσεις τουλάχιστον, καθόλου κοντά δεν είναι στη Χάγη. Καλά σας τα λέω. Νομίζω ότι είναι μια πλήρως εσφαλμένη απόφαση του Συμβουλίου. Θα θέλαμε όμως ε, να ψηφίσουμε επί της ε, συμβαστικής πρότασης για να δούμε αν θα καταφέρουμε να επηρεάσουμε το τελικό αποτέλεσμα. Uh, just a brief response to Mr. Duff. Να απαντήσω σύντομα στον κύριο Νταφ. Υπάρχει πολύ καλή ε, επικοινωνία ρωματοφορών μεταξύ Σχίπχολ και Βουδαπέστη. Επομένω, το γεωγραφικό σκέλος αυτή τη στιγμή δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία. Σημειώνω την παρατήρησή σα. Α, έφτασε όμω και η συγκήτρια, βλέπω. Φαντάζομαι ότι ε, κατάφερε να φύγει νωρίτερα από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, στην οποία ήταν. Κυρία Τέιν, θα ξεκινούσαμε την ψηφοφορία για την έκθεσή σας. Δεν ξέρω αν θέλετε να πάρετε το λόγο. Όχι, νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να ψηφίσουμε. Λοιπόν, ψηφίζουμε καταρχάς. Συμφωνείτε, καταρχάς, πείτε μου αν συμφωνείτε με αυτό που θα σας πω τώρα. Θα μπορούσαμε να ψηφίσουμε τις τροπολογίες από την 1 μέχρι την 4 μαζί. Να τις ψηφίσουμε από κοινού. Ουσιαστικά δύο σελίδες τροπολογιών να τις ψηφίσουμε από κοινού. Αν συμφωνεί η συγκήτρια που βλέπω ότι συμφωνεί, τότε μπορούμε να ψηφίσουμε από κοινού τις τροπολογίες αυτές. Ψηφίζουμε λοιπόν τις τροπολογίες οι οποίες εμφανίζονται στον κατάλογο ψηφοφοριών από την 1 έως την 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται ομόφωνα. Συμβαστική Α, όπου έχουμε και την ε, αναφορά για τις κοντινές αυτές έδρας. Δεν νομίζω πάντως ότι ο κύριος Ντάφ ζήτησε να γίνει κάποια τροποποίηση, μα ζήτησε να παραμείνει το κείμενο ως έχει. Ψηφίσουμε λοιπόν τη συμβαστική α, υπέρ. Κατά. Δύο ψήφοι αποχές, εγκρίνεται. Τρεις ψήφοι κατά. Οι υπόλοιπε τώρα τροπολογίες, μάλλον έχουμε τη συμβαστική Β. Έχουμε μάλλον την τροπολογία 6 λέει ο πρόεδρο της εισηγήτρια, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία B. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται ομόφωνα καταπίπτουν οι 22 και οι 7. Νομίζω ότι οι τελευταίες τρεις τροπολογίες, 8, 57 και 58, μπορούν να τις ψηφίσουμε από κοινού υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται, ομόφωνα. τελική ψηφοφορία για το σύνολο του κειμένου ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία. Δεν έχετε την κάρτα σας. Θα σας προσθέσουμε μετά. Άρτη ψηφοφορία. Στην οθόνη βλέπουμε ότι έχουμε τρεις επιπλέον ψήφους από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. τρεις επιπλέον ψήφοι από το ΕΛΚΑ. Πρέπει λοιπόν να αφαιρέσουμε αυτές τις τρεις επιπλέον ψήφους. Και να προσθέσουμε όμως και την ψήφο της κυρίας Σατέιν. Ένας ακόμα επιπλέον εμφανίστε εδώ στην οθόνη μου, από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα πάντα να βγάλουμε. Έχουμε πάντως μία ψήφο επιπλέον ακόμα. Κανείς δεν αισθάνεται εδώ πέρα περίτως, προκειμένου να αποσύρει την ψήφο του. αντικαταστήσουμε τον πρόεδρο. Πολύ ωραία πρόταση, μάλιστα. Μάλιστα, πολύ ωραία. Το λύσαμε το πρόβλημα. 26 ψηφίσαντες, ουδής κατά, καμία αποχή, εγκρίνεται λοιπόν ομόφωνα. Συγχαρητήρια κυρία Τέιν. Περνάμε τώρα στην έκθεση Τρασκόφσκι για τη διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά ναι, ναι, ένα λεπτό. Σχετικά με τη συνεργασία σε θέματα προπολογισμού και χρηστής διαχείρισης. Νομίζω ότι ο κύριος Γκουαλτιέρη θέλει το λόγο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι ήταν χρήσιμο να αποσαφηνίσουμε εδώ πέρα ότι για τη δική μου την πολιτική ομάδα αλλά και για όλη την Επιτροπή η έγκριση της έκθεσης αυτής στην Επιτροπή μας αποτελεί ένα μόνο πρώτο βήμα. Εμείς θεωρούμε ότι η τελική ψηφοφορία στην Ολομέλεια θα εξαρτηθεί τελικά από την θετική έκβαση όλων των διαπραγματεύσεων για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ήθελα απλώ να κάνω τη διευκρίνηση αυτή, έτσι ώστε να μην ερμηνευθεί η σημερινή ψηφοφορία ως πράσινο φως μιας συμφωνίας η οποία ακόμα εκκρεμεί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρατήρηση σας αυτή και εγώ αυτό είχα πει αρχικά όταν παρουσίαζα την ημερήσια διάταξη, λέει ο Πρόεδρος, ο κύριος Τάφα. Ναι, εκ μέρους της ομάδας των φιλελευθέρων. Συμφωνώ με τις παρατηρήσεις του κύριου Βατιέρη. Ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις μεταξύ όλων των επιτροπών και του Συμβουλίου επί αυτού του ζητήματος. Παρότι είμαστε διατεθειμένοι να προχωρήσουμε και έτοιμοι να προχωρήσουμε στην Επιτροπή, θα πρέπει και πάλι να το εξετάσουμε εκ νέου στο Στρασβούργο για την Ολομέλεια, όταν θα έχουν ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Και θα ήθελα να ρωτήσω τον εισηγητή. Συμφωνείτε υπό τον ε, πρώτο συμβασμό; αντί να πούμε welcomes, χαιρετίζουμε, δηλαδή επικροτούμε την πολιτική απόφαση, να πούμε μόνο note. Αντί για welcome να πούμε note, λοιπόν, για το πολιτές νομικό πλαίσιο, γιατί δεν θεωρώ ότι πρόκειται και για μια ιδιαίτερα λαμπρή στιγμή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο άφησε την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς τους πόρους που χρειάζεται για να επιτύχει πλήρως και να εκπληρώσει τις ε, πολιτικές ε, και νομικές της υποχρεώσεις. Συμφωνείτε κύριε Ταρκόφσκι. Ο κύριος Λαμασούρ μάλλον πρώτος. Euh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, για αυτά που είπε ο κύριος Βαλτιέρη, αυτό αντιστοιχεί απολύτως με την απόφαση της διάσκεψης προέδρων των ομάδων την προηγούμενη εβδομάδα, που επιβεβαίωσε ότι η τελική ψηφοφορία για την διοργανική συμφωνία και τον κανονισμό που λέει του δημοσιονομικού πλαισίου θα γίνει κατά τη δεύτερη ε, σύνοδο ολομέλεια ε, στις 23 Οκτωβρίου δηλαδή, αρκεί να έχουν επιληθεί δύο κατηγορίες προβλημάτων που ε, την χάνουν διαπραγματεύσεων αυτή τη στιγμή. Έχουμε και κάποιες ε, νομοθετικά προβλήματα και άλλες θέματα που αποτελούν αντικείμενο τεμερών διαλόγων. Η σημερινή ψηφοφορία έχει ως στόχο να καταστήσει πιθανή και δυνατή τη ψηφοφορία στις 23. Εάν δεν τη ψηφίσουμε σήμερα, τότε δεν μπορούμε να πάμε ε, στην Ολομέλεια στις 23 και αναβάλλεται για ένα μήνα ακόμα. Η διάσκεψη των Προέδρων είχε πολύ ξεκάθαρη θέση να τεθεί, ε, να θέσει υποπίεση το Συμβούλιο. Και μετά βλέπουμε, όπως είπαν και οι συνάδελφοι, αν ε, πληρούνται οι προϋποθέσεις. Και η διάσκεψη των Προέδρων θα το αποφασίσει. Για την προφορική τροπολογία που πρότεινε ο συνάδελφος Νταφ, Ω πρόεδρος τη Επιτροπής Προπολογισμών και με τον πρόεδρο Σούλτ, ε, που είναι ο βασικό διαπραγματευτή επί το περιεχομένου συμφωνίας είμαι αντίθετος. Εδώ δεν λέμε ότι σημειώνουμε note, πρέπει να πούμε αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε. Και επιμένω να διατηρήσουμε το welcomes, επικρατούμε, χαιρετίζουμε, γιατί αλλιώς σημαίνει ότι η ΆΜΚΟ διαφωνεί ε, ή τέλο πάντων δεν συμφωνεί με τι διαπραγματεύσει. Επομένω ε, δεν μπορώ να συμφωνήσω με αυτή την πρόταση. Ο κύριο Νταφ, ε, ναι βεβαίω και εκτιμώ τη θέση του Προέδρου τη Επιτροπή Προπολογισμού. Αν ε, δεν συμφωνεί με το note, μήπως συμφωνεί με το accepts, αποδέχεται το αποτέλεσμα. Δηλαδή, δεν επικροτούμε και δεν χαιρόμαστε και ιδιαίτερα, δεν πετάμε τη σκούφια μας. Ε, εντάξει. Λοιπόν. non ci sono allora a Λοιπόν, αν δεν υπάρχουν λοιπόν αντιρρήσεις για την προφορική αυτή τροπολογία, η οποία τροποποιεί την συμβαστική τροπολογία Α. Εφόσον λοιπόν δεν υπάρχουν ε, αντιρρήσεις, συμβαστική Α υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Καλύπτονται κατά αυτόν τον τρόπο οι τροπολογίες 1 και 4 και μπορούμε να περάσουμε τώρα στην βασική Β υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Και καλύπτονται έτσι τροπολογίες 5 και 2 της Επιτροπής Τροπολογισμών. Μπορούμε τώρα να ψηφίσουμε τη συμβαστική τροπολογία C υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Καλύπτονται κατά αυτόν τον τρόπο τροπολογίε 6 και τροπολογία 3 τη επιτροπή Προπολογισμών. Αποσύρεται η τροπολογία 7. Ψηφίζουμε την τροπολογία 4 τη επιτροπή Προπολογισμών. Υπέρ. Υπέρ για την τροπολογία 4. Κατά. Τροπολογία 5 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8, με συγχωρείτε, 6 της Επιτροπής Προπολογισμών. Υπέρ. Κατά. αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8 του κυρίου Έφνερ. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 9. Υπέρ. κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 1, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 2, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Περνάμε στην τελική ψηφοφορία για την έκθεση αυτή. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Έχουμε μία επιπλέον ψήφο από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Εντάξει, διορθώθηκε το πρόβλημα. Άρθη ψηφοφορία. Πέρας. 21 υπέρ, 5 κατά, καμία αποχή.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 Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε κανονικά ε, μέλη και αναπληρωματικά μέλη, τα οποία όμως συμμετέχουν κανονικά στις εργασίες της Επιτροπής. Ε, γι' αυτό έγινε αυτό ε, που παρατηρήσατε. Θα προσπαθήσουμε όμως. Όχι, δεν αναφερόμουν στα μέλη και τα αναπληρωματικά μέλη. Αναφερόμουν σε μέλη που δεν, δεν ψηφίζουν, ψήφισαν. Γι' αυτό το είπα. that... Uh, να διευκρινίσω ότι κάθε πολιτική ομάδα θα πρέπει να ακολουθεί τους ε, κανόνες των ψηφοφοριών. Όμως η πολιτική ομάδα αποφασίζει ποιος θα παρευρεθεί στην ψηφοφορία. Μπορεί να υπάρξει υποκατάσταση μέλους εάν αυτό είναι απαραίτητο. Ε, οι υπεύθυνοι κάθε πολιτικής ομάδας σας διασφαλίσουν ότι ε, θα ψηφίζουν αυτοί οι οποίοι πρέπει να ψηφίσουν ε, για να μην καταλήγουμε με επιπλέον τελικά ψήφου. Ενδεχομένω οι επικεφαλεί λοιπόν των πολιτικών ομάδων να πρέπει να επιβάλλουν λίγο την τάξη. Ας ψηφίσουμε όμως τώρα την έκθεση Λαμασούρ, να αλλάξουμε δηλαδή τη σειρά που προβλέπετε, πριν ψηφίσουμε την έκθεση Φόξ και Ο κύριος Λαμασούρ μου ζήτησε να ψηφίσουμε πρώτα τη δική του την έκθεση δυνατών, γιατί θα πρέπει να αποχωρήσει πριν τη λήξη της συνεδρίασης. Γι' αυτό το λόγο περνάμε ευθύ αμέσω στην ψηφορία της έκθεσης του κυρίου Λαμασούρ, όσον αφορά τις σχέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τα θεσμικά όργανα που εκπροσωπούν τις ε, εθνικές κυβερνήσεις. Νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε αμέσως λοιπόν στην ψηφοφορία αυτής της έκθεσης. Θέλετε να πάρετε το λόγο κύριε Λαμασούρ, παρακαλώ. Euh, να σας ευχαριστήσω καταρχήν κύριε Πρόεδρε καθώς και τους συναδέλφους. Επίσης θα ήθελα να σας πω ότι μετά από πρόσφατες επαφές με τους συναδέλφους έχω τέσσερις προφορικές τροπολογίες που βελτιώνουν τις συμβιβαστικέ. Η μία στο D, νέα παράγραφος 8, Επίσης, άλλη τροπολογία για την συμβιβαστική F, αλλά και στην θέση προς αντικατάσταση της τροπολογίας 9 και 13. Μπορείτε να μας να, τα ξαναπείτε αυτά κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, να μας το τονίσετε, δηλαδή όταν φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Υπάρχουν άλλοι που θέλουν να πάρουν το λόγο. Διαφορετικά, ξεκινάμε την ψηφοφορία. Ψηφίζουμε τη συμβαστική α. Μάλλον την τροπολογία 27 πρώτα. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Περνάμε στην συμβαστική τροπολογία α, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Πράγμα σημαίνει ότι περνάμε στη συμβαστική B. Ο κύριος Ντάφ το λόγο. Εγώ είχα ζητήσει να γίνει ψηφοφορία κατά τμήματα στο, για το τελικό τμήμα αυτής της συμβιβαστικής Ξεκινώντας με τη φράση οι συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου δεν θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της εβδομάδας της Ολομέλειας. Θα ήθελα λοιπόν, επειδή είμαι κατά αυτού του τμήματος, αλλά συμφωνώ με το πρώτο τμήμα αυτής της συμβαστικής τροπολογίας, να ζητήσω ψηφοφορία κατά τμήματα. Est-ce que j'aurai le droit de faire un amendement oral pour essayer d'aller au-devant de Andrew Alors, si oui, l'amendement consisterait à dire, à remplacer euh, not, euh, not take place during the plenary session weeks Uh, at the end of the το τέλος εβδομάδας Ολομέλεια. Δηλαδή, ο κύριος Νταφ, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν θα πρέπει να συνεδριάζει στο τέλος των κοινοβουλευτικών των εβδομάδων κοινοβουλευτικών συνεδριάσεων. Αυτό συμβαίνει συχνά το Συμβούλιο συνεδριάζει την Πέμπτη και την Παρασκευή των εβδομάδων της Ολομέλειας. Άρα δεν μπορεί να έρθει ο πρόεδρος κατά τη διάρκεια της εβδομάδας της Ολομέλειας παρά μόνο ένα μήνα αργότερα. Γιατί αν συνεδρίαζαν παραδείγματος χάρη Δευτέρα και Τρίτη θα μπορούσαν να έρθουν Πέμπτη και Παρασκευή να μας παρουσιάσουν τα αποτελέσματα του Συμβουλίου. Ο κύριος Νταφ. Το πρόβλημα είναι ότι αν λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της εβδομάδας της Ολομέλειας δεν είναι σε θέση ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου να πάρει το λόγο στο Συμβούλιο με μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ούτε την Πέμπτη και την Παρασκευή δηλαδή, γιατί αναγκάζεται ο Πρόεδρος να πάρει το λόγο χωρίς να έχει την απόφαση μιας, ε, της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου. Ο κύριος Γκουαλτιέρη, από ό,τι κατάλαβε υπάρχουν δύο αντιτιθέμενες απόψεις, άρα το καλύτερο είναι να ψηφίσουμε. Νομίζω ότι έχουμε μία προφορική τροπολογία, η οποία δεν συνάδει, μάλλον λέει το αντίθετο από αυτό το οποίο λέει ο Άντριου. Ο κύριος Λαμασούρ προτείνει να μην γίνεται το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μετά την Σύνοδο Λομέλειας, ενώ σύμφωνο, σύμφωνα με τον Άντριο αυτή θα ήταν η καλύτερη στιγμή. Επομένως καταλαβαίνετε ότι έχουμε δύο αντιτιθέμενες απόψεις, το καλύτερο να ψηφίσουμε και να δούμε ποια θα είναι η έκβαση. Εμείς υποστηρίζουμε πάντως την πρόταση του κυρίου Λαμασούρ. Κύριε, Λαμασούρ, ε, κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε, αποσύρω την προφορική μου τροπολογία και σας προτείνω να κάνετε αυτό το οποίο σας ζήτησε ο κύριος Δάφτη, δηλαδή χωριστή ψηφοφορία, ψηφοφορία κατά τμήματα όσον αφορά την τελευταία αυτή φράση. Εγώ θα ψηφίσω υπέρ της τελευταίας φράσης, γιατί κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να εξυπηρετήσουμε και την άποψη της κυρίας για την Νομίζω ότι και οι δύο απόψεις είναι σωστές. Στη μία περίπτωση ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μπορεί να είναι παρόν στο Στρασβούργο στην Ολομέλεια, ενώ σύμφωνα με την άλλη άποψη ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου θα έχει εντολή για να πηγαίνει και να μιλάει σε συνόδους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Και τα δύο είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και η εντολή που δίνουμε εμείς στον πρόεδρό μας για να πηγαίνει στο Συμβούλιο, αλλά και να μπορούμε να ακούμε τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στι Ολομέλειες του Στρασβούργου. Δεν ξέρω πώς θα διευθετήσουμε αυτό τώρα με τις τροπολογίες, πάντως θεωρώ ότι οι δύο προσεγγίσεις είναι πολύ σωστές και απαραίτητες. Και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πρέπει να έρχεται στο Κοινοβούλιο, αλλά και ο δικός μας ο πρόεδρος πρέπει να πηγαίνει και να μιλάει και να έχει μια συγκεκριμένη εντολή από εμά στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Πρέπει να καταφέρουμε να διευθετήσουμε, πιστεύω, και τις δύο απόψεις στο κείμενο. Πρόεδρος, κοιτάξτε, ουσιαστικά μας λέτε ότι είστε υπέρ του να γίνονται την Πέμπτη και την Παρασκευή το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ο κύριος Λαμασούρ όμως απέσυρε τώρα την προφορική του τροπολογία και μας ζήτησε να κάνουμε κατά τμήματα ψηφοφορία σύμφωνα με τα όσα ζήτησε ο κύριος Ντάφα. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό μπορούμε να κάνουμε. Ψηφίσουμε το πρώτο τμήμα της συμβαστικής τροπολογίας B. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα της συμβαστικής τροπολογίας B υπέρ κατά. Εγκρίνεται. Καλύπτονται από τη συμβαστική 31 και 32, ψηφίσουμε την 33 του κ. Ντάφ υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 34 του κυρίου Χέφνερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία C υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται καλύπτονται κατά αυτόν τον τρόπο οι 35 και ψηφίζουμε την 36 για την παράγραφο 6 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Αποχές μάλλον. Απορρίπτεται. Τροπολογία 37 Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 37 της κυρίας Γιαννάκου. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Ένας επιπλέον ακόμα. 13 υπέρ 13 κατά απορρίπτεται Τροπολογία ψηφίσαμε την 37, περνάμε στην 38 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 39. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία D. Κύριε Λαμασούρ, το λόγο. Merci, le Président. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Για την συμβαστική D υπάρχει αίτημα για κατατμήματα ψηφοφορία. Για το πρώτο τμήμα λοιπόν έχω μια προφορική τροπολογία σε σχέση με τη συμβαστική τροπολογία που είχα προετοιμάσει για να λάβω υπόψη μου την ε, τροπολογία Γκουρμάη και αφού μίλησα και με τον κύριο Κουαλτιέρη, ο οποίος ήθελε να γίνει πιο σαφής η διατύπωση του κειμένου όσον αφορά την υποχρέωση του Συμβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να συμφωνήσουν ε, όσον αφορά τον ε, διορισμό του Προέδρου της Επιτροπής. Θεωρεί λοιπόν ο συνάδελφος Γουαλτιάρη ότι η δική μου διατύπωση δεν είναι αρκετά ε, σαφής και ακριβής. Σας προτείνω λοιπόν να διατυπώσουμε ως εξής το πρώτο τμήμα αυτού, αυτής της νέας παραγράφου 8. Καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να γνωστοποιήσει με σαφή τρόπο πριν την αρχή των ευρωπαϊκών ε, της προεκλογικής περίοδου των ευρωπαϊκών εκλογών Όσον αφορά το Συμβούλιο, πώς προτίθεται να σεβαστεί την άποψη των Ευρωπαίων πολιτών όσον αφορά το διορισμό του Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βάσει του άρθρου 17 παράγραφος 7 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επαναλαμβάνω, άρθρο 17 παράγραφος 7 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια των διαβουλεύσεων μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με το άρθρο αυτό το οποίο θα προσαρτηθεί. Δηλαδή ζητούμε από το Συμβούλιο να διευκρινίσει πως το Συμβούλιο προτίθεται να ε, σεβαστεί την άποψη των Ευρωπαίων Πολίτων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εδώ γίνεται μια σαφής μνήμα στο άρθρο 17 παράγραφο 7 των συνθήκων. Και κατόπιν προτείνω να ψηφίσουμε το δεύτερο τμήμα. Εδώ πρόκειται για το πρώτο τμήμα. Πρόεδρος. Μάλιστα, ακούσατε πολύ καλά τα όσα μας είπε ο κύριος Λαμασούρ με απόλυτη σαφήνεια. Ψηφίζουμε λοιπόν το πρώτο τμήμα της συμβαστικής D κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα της συμβαστικής D υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση για το δεύτερο τμήμα. Άρτη ψηφοφορία. Πάλι μία ψήφος επιπλέον. Θα θυσιαστώ εγώ. Ελπίζω να μην αλλάξει η έκβαση της ψηφοφορίας. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. 15 υπέρ, 10 κατά, καμία αποχή. Εγκρίνεται και το δεύτερο τμήμα της συμβαστικής τροπολογίας D. Περνάμε τώρα Τροπολογία 41. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 42. Υπέρ. κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται ηλεκτρονική επαλήθευση πολύ ωραία ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την τροπολογία 42 Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εννέα υπέρ, 17 κατά, καμία αποχή. Απορρίπτεται. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 43. Υπέρ. Κατά. Αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση, άρτη ψηφοφορία. Πέρας. 10 υπέρ, 16 κατά, καμία αποχή, απορρίπτεται. Περνάμε τώρα στις αιτιολογικές αναφορές, τροπολογία 1 υπέρ, κατά αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά μπορούμε να επαληθεύσουμε και ηλεκτρονικά άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. 16 υπέρ, 10 κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 2 του κύριου Έφνερ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 του κυρίου Ντάφ υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 4. Διορθώνει ο πρόεδρος. Συμβαστική τροπολογία E υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Άρα, καλύπτονται οι υπόλοιπες τροπολογίες μέχρι την 41. Pongo in votazione allora l'emendamento 7. Τροπολογία 7. Υπέρ. Διευκρινίζει ο πρόεδρο ότι υπάρχουν αρκετά τμήματα στην τροπολογία 7, τρία συγκεκριμένα τμήματα. Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα τη τροπολογία 7 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα τη τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 8 υπέρ κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 9 Προφορική τροπολογία από την εισηγητή υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Allora, l'emendamento 10 va votato in tre parti. Sì. Τροπολογία 10 se tre tmimata, proto tmima, iper. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 13. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την τροπολογία 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. 12 υπέρ, 14 κατά, καμία αποχή, απορρίπτεται. Τροπολογία 16. Καταπίπτει. Ναι, όντως, καταπίπτει 16. Περνάμε στη συμβαστική τροπολογία F. Ο κύριος Λαμασούρ. Oui, merci, monsieur le président. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Προτείνω εδώ μια προφορική τροπολογία στο τέλος αυτής της συμβιβαστικής τροπολογίας F γιατί ο κύριος Κουαλτιέρη μου υπενθύμησε ότι αυτό που γράφουμε στο κείμενο αυτής της συμβαστικής τροπολογίας είναι λίγο επικριτικό προς τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, τον αποδυναμώνει. Προτείνω λοιπόν μια νέα σύνταξη για τις δύο τελευταίες σειρές αυτής της τροπολογίας, μετά δηλαδή την ε, ανοτελιά εκεί που λέει ότι το Συμβούλιο παίζει ένα ρόλο χωρίς ουσιαστική σημασία, παρόλη την σημασία η παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Προέδρου μάλλον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην έναρξη των συμβουλίων δεν είναι επαρκής διαδικασία. Δηλαδή, με αυτή την νέα διατύπωση δεν ε, επικρίνουμε τον πρόεδρο. Λέμε ότι είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που κάνει, αλλά δεν αρκεί. Εξάλλου αν αρκούσε, αν ήταν επαρκής η διαδικασία αυτή, δεν θα κάναμε καθόλου αυτή την έκθεση, αυτή την πρόταση. Προτείνω λοιπόν να ψηφίσουμε το κείμενο της συμβαστικής τροπολογίας με την τροπολογία αυτής της δύο τελευταίες σειρές. Πρόεδρος. Δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, άρα μπορούμε να ψηφίσουμε τη συμβαστική F με την προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 17 σε κατατμήματα. Ecco sì, esatto. Andiamo così all'emendamento 19. Περνάμε μάλλον στην τροπολογία 19 του κύριου Λάινεν υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά μπορούμε να επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Λοιπόν, ηλεκτρονική επαλήθευση για τροπολογία 19. Άρτε ψηφοφορία. Πέρας. 10 υπέρ, 15 κατά, απορρίπτεται. Και καμία εποχή. Τροπολογία 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται νομίζω. Ναι, εγκρίνεται. Τροπολογία 21 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 22 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 23 υπέρ. Κατά. Αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση. Για την τροπολογία 23. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Το υπέρ, 17 κατά, καμία αποχή. Απορρίπτεται. Τροπολογία 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 25 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 26 υπέρ. Κατά αποχές, η ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 26 του κυρίου Λάινεν, άρτη ψηφοφορία. Πέρας. 11 υπέρ, 15 κατά, απορρίπτεται. Ψηφίσουμε τώρα το σύνολο της πρώτας ψηφίσματος. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με 22 ψήφους υπέρ, 4 κατά, καμία αποχή. Σας ευχαριστώ όλους και να ευχαριστήσω βέβαια τον εισηγητή μας τον κύριο Λαμασούρ. Όχι μόνο για τη σημερινή του εργασία, αλλά για την εργασία που έχει κάνει όλο το τελευταίο διάστημα. Κύριος Λαμασούρ, σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Passiamo al voto. Ψηφίζουμε τώρα την έκθεση Fox και Έφνερ για το καθορισμό της έδρας των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Έφνερ, έχετε τον λόγο. Could I just have a short before we start voting?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 γιατί είναι προφανώς ότι δεν υπάρχει κάποια σκόπιμη παρατυπία, αλλά υπάρχει σύγχυση. Μάλιστα. Μία προκαταρκτική επαλήθευση μπορούμε να κάνουμε αν θέλετε. Δηλαδή επικεφαλής των πολιτικών ομάδων να ξεκαθαρίσουν αυτή τη στιγμή ποιος ψηφίζει και ποιος όχι. Ξεκινάμε με το ΕΛΚ. Κοιτάξτε, εγώ δεν συμμετείχα πολλές φορές ε, στις προφορίες γιατί πάντα έβλεπα ότι υπήρχε μία επιπλέον ψήφος από το ΕΛΚ. Καταλαβαίνω βέβαια τόσο, λέει ο κύριος Σέφνερ, έχει απόλυτο δίκιο στις παρατηρήσεις του. Εγώ μπορώ να συνεχίζω να μην ψηφίζω όπως έκανα. Ο κύριος Ταρκόφσκι. Ε, Κοιτάξτε, υπάρχουν δέκα ψήφοι. Όλα τα πλήρη μέλη έχουν προτεραιότητα και κατόπιν εάν λείπουν κάποια πλήρη μέλη, συμπληρώνονται με τα αναλπιρωματικά. Ε, Αυτό σημαίνει ότι βεβαίως και μπορεί να ψηφίσει ο πρόεδρος. Compreso me Εμού νομίζω ότι είμαστε 12 από το ΕΛΚ. Πρόεδρε, το θέμα είναι τι γίνεται με εσά, γιατί θέλετε να ψηφίσετε αν κατάλαβαμε καλά. Δηλαδή να φύγει ένα από τα αναπληρωματικά μα μέλη. Εντάξει. Κοιτάξτε, εγώ δεν είπα σε κανέναν ότι θέλω, δεν θέλω να ψηφίσω. Αλλά καθότι είμαι πρόεδρος, πρέπει να είμαι και κάπως ε, ανεξάρτητος, ως το δυνατόν περισσότερο. Επομένως, ε, δέχομαι να μην ψηφίσω εγώ. Αρμόζει περισσότερο με το ρόλο μου. Λαμασούρ και Μπλάνκοβιτς δεν θα ψηφίσουν. Ο κύριος Λαμασούρ δεν θα ψηφίσει. Allora, il Presidente del Gruppo ha fatto il calcolo di... Λοιπόν, στους 10 ποιοι συμμετέχουν από το ΕΛΚ αυτή τη στιγμή, ποιοι μπορούν να ψηφίσουν. Τα μέλη του ΕΛΚ που θα ψηφίσουν αυτή τη φορά μπορούν να σηκώσουν το χέρι παρακαλώ για να είμαστε σίγουροι. Γιατί συνέχεια παίρνω λανθασμένες πληροφορίες. 10. We are fine. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ωραία, ευχαριστούμε. Nice to see Πρόεδρε, χαίρομαι που είναι τόσο πολλοί οι Γάλλοι συνάδελφοι στην ΑΜΚΟ. Ελπίζω και να έρθουν, ξαναέρθουν στις συζητήσεις μας όταν δεν θα συζητούμε το θέμα του Στρασβούργου. Λοιπόν, ανάλογος έλεγχος πρέπει να γίνει και με τις άλλες πολιτικές ομάδες. Δεν νομίζω Πολύ ωραία. Περνάμε λοιπόν στην ψηφοφορία της έκθεσης ε, Έφνερ και Φόξ. Ξεκινάμε με την τροπολογία 85. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 86. Υπέρ. Καλύτερα να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για την τροπολογία 86 της κυρίας Λεγκρίπ. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 10 υπέρ, 16 κατά. Καμία αποχή. Τροπολογία 87. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρτη ψοφορία Πέρας. 9 υπέρ, 17 κατά, καμία αποχή απορρίπτεται. Τροπολογία 88 υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 89 υπέρ, κατά αποχές. Καλύτερα να ψηφίσουμε και ηλεκτρονικά για αυτήν την τροπολογία, άρτη ψηφοφορία. Πέρας. 11 υπέρ, 15 κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 90. Υπέρ. κατά αποχές εγκρίνεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση μάλλον, άρθρη ψηφοφορία. Πέρας. 12 υπέρ και 12 κατά, μία αποχή, άρα απορρίπτεται. Τροπολογία 91 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την 91. Πέρας. 10 υπέρ, 15 κατά μία αποχή. Απορρίπτεται. 92 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με 15 υπέρ και 10 κατά μία αποχή. Υπολογή υπαριθμών 1 της Επιτροπής Αναφορών. Ψηφίζουμε μόνο το δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική ψηφοφορία τώρα, πάλι για την υπαριθμόν 1 της Επιτροπής Αναφορών, άρθρη ψηφοφορία. Πέρας. 14 υπέρ, 11 κατά, μία αποχή εγκρίνεται. Τροπολογία 93. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 94. Υπέρ. Κατά ηλεκτρονική επαλήθευση, άρθρη ψηφοφορία. Πέρας. 11 υπέρ, 15 κατά, καμία αποχή. Απορρίπτεται. 95 υπέρ. Κατά. Αποχές. Η ηλεκτρονική επαλήθευση και για την 95. Άρτε ψηφοφορία. Πέρας. 11 υπέρ, 15 κατά, καμία αποχή, απορρίπτεται. 96. Ηλεκτρονική επαλήθευση, αμέσως. Υπέ, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. 11 υπέρ, 15 κατά, καμία αποχή, απορρίπτεται. 97. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. 10 υπέρ, 15 κατά. Απορρίπτεται. 98. Υπέρ. Με συγχωρείται ο πρόεδρος. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. 24 υπέρ, μία ψήφος κατά, μία αποχή. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε λοιπόν στην τροπολογία 105. του κυρίου Μπουλάν. Υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται. Τροπολογία υπαριθμών 4 της Επιτροπής Αναφορών υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 106 της κυρίας Λεγκρίπ υπέρ κατά αποχές Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά ας επαληθεψουμε ηλεκτρονικά. Άρτη ψηφοφορία. Την 106 ψηφίζουμε, της κυρίας Λεγκρίπ. Πέρας λοιπόν, 11 υπέρ, 15 κατά, απορρίπτεται. 107 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 108 του κυρίου Μπελιέ, της κυρίας Μπελιέ, υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. 109 του κύριου Νταφ έχει αποσυρθεί, 110 του κύριου Μπουλά, καταπίπτει, Απολογία 111 υπέρ κατά αποχές Ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά άρθρη ψηφοφορία πέρας 13 υπέρ, 10 κατά, 3 αποχές εγκρίνεται. 112. Γκυγιόμ και Τροτμάν. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 113 του κύριου Μπουλάν. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται.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 121 υπέρ, κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 122 και έχουμε και προφορική τροπολογία εδώ. Μπορούμε πάντως να την ψηφίσουμε υπέρ για την 122, κατά, αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση, νομίζω πάντως ότι εγκρίνεται άρτη ψηφοφορία. Πέρας. 14 υπέρ, 12 κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 3 της Επιτροπής Αναφορών, η οποία όμως καλύπτεται από την τροπολογία 122, την οποία την έχουμε εγκρίνει, άρα δεν ψηφίζουμε την 3. Νομίζω ότι και η τροπολογία υπαριθμών 1 της Επιτροπής Τροπολογισμών έχει και αυτή καλυφθεί από προηγούμενες τροπολογίες που έχουν εγκριθεί. Το ίδιο ισχύει, μάλλον όχι. Τροπολογία υπαριθμών 2 της Επιτροπής Προπολογισμών. Υπέρ. Κατά. Η ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρθει ψηφοφορία. Πέρας. Τρεις ψήφοι υπέρ, 23 κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5 της Επιτροπής Αναφορών. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 6 της Επιτροπής Αναφορών υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 6 της Επιτροπής Αναφορών, άρθρο ψηφοφορία, πέρας. Εγκρίνεται με 16 ψήφους υπέρ, 9 ψήφους κατά και 3 αποχές. Νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε ηλεκτρονικά από εδώ και πέρα. 123 του κυρίου Μακμίλαν Σκοτ. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Τρεις ψήφοι πέρ, 22 κατά, μία αποχή. Απορρίπτεται. 124 Μακμίλαν Σκοτ. Ηλεκτρονικά και πάλι. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Νομίζω ότι διανατάσσεως θα ήταν ξεκάθαρο το αποτέλεσμα, απορρίπτεται. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 1, διανατάσσεως αυτή τη φορά υπέρ, κατά. ηλεκτρονική επαλήθευση όμως και πάλι χρειαζόμαστε, άρχεται ψηφοφορία για την τροπολογία περιθμών 1. Πέρας. 11 υπέρ, 14 κατά, τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρτη ψηφοφορία. Εκείουσα βοτατσιόνε. Πέρας. Απορρίπτεται. Τρία. Υπέρ. Με ο χειρός. Κατά. Μου φαίνεται ότι υπάρχει λουψία. Απορρίπτεται. πέντε Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική J. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Αυτό σημαίνει ότι ψηφίζουμε την 7 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 8 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 9 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Β, συμβιβαστική Β, Β, υπέρ. Κατά. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Αρχή. Πέρας. Υπέρ με εφορά δύο ψήφων. Ε, εγκρίνεται, συγγνώμη. Και τώρα πάμε στη συμβαστική α. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Α. Συμβαστική α. Αρχή της ψηφοφορίας. Πέρας. Με ομοφωνία εγκρίθηκε και περνάμε στη 14. Μακμίλαν. Υπέρ. κατά εγκρίνεται. Σίγουρα εγκρίνεται. Και τώρα πάμε στη 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 16. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται σίγουρα εγκρίνεται 19 προφορική τροπολογία Βίλαντ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 20. Όχι, 21 εγκρίθηκε, άρα καταπίπτει. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 23 υπέρ. Κατά. Αποχές Ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 23 αρχή της ψηφοφορίας. Πέρας. 12 υπέρ, 14 κατά. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 26 κατά αποχές απορρίπτεται 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται περνάμε συμβαστική C υπέρ ηλεκτρονική ψηφοφορία. Συμβιβαστική C. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρας. Εγκρίνεται. Αυτό σημαίνει ότι περνάμε στη συμβαστική D. Υπέρ αποχές εγκρίνεται. Και τώρα πάμε στην 36 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική ψηφοφορία. Αρχή της ψηφοφορίας, τέλος. απορρίπτεται. Και τώρα περνάμε στην προφορική τροπολογία την, του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 37 όχι όχι Έχω μία προφορική τροπολογία. Εκεί που λέει 736 ε, μέλη, θα προσθέσουμε τη λέξη currently, γιατί αυτό μπορεί να αλλάξει. Θέλεις να προσθέσεις δηλαδή τη λέξη currently, προς το παρόν. Ο εισηγητής... Αν μπορούν το δεχτούν οι εισηγητές, νομίζω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν υπάρχει λόγος τώρα να επανλάβουμε όλη την ψηφοφορία. Συμφωνείτε λοιπόν με αυτή τη νέα προφορική τροπολογία. Νομίζω ότι συμφωνούστε το σε άλλους όλοι κατά αποχές, άρα εγκρίνεται με αυτή την διευκρινιστική προφορική τροπολογία. 37 υπέρ. Κατά. 37 ψηφίζουμε. Καταπίπτει. συγγνώμη, ελέγχουμε. Κύριε Ντάφου, λέτε ότι καταπίπτει γιατί είναι αντίθετη με κάποια άλλη. Α, ναι, ναι, ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο, όπως πάντα έχει δίκιο ο κύριος Ντάφου. Η 37 καταπίπτει. Η 38. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται 39 υπέρ. κατά αποχές απορρίπτεται 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ένα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται α ηλεκτρονική Ψηφοφορία για την 41. Αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Εγκρίνεται. Είχα δίκιο. Ωραία. Και τώρα εγκρίθηκε η 41. Η 42 καταπίπτει και περνάμε 43 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 44 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 45 45 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 47 υπέρ κατά ηλεκτρονική ψηφοφορία. 47. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται για μία ψήφο. 13-12. 48 υπέρ. να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για την 48. Αρχή της ψηφοφορίας. Πέρας. Απορρίπτεται. 49. Αρχή της ψηφοφορίας. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική ε. Ψηφίζουμε υπέρ. Ηλεκτρονικά. Αρχή της ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. 61. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Αρχή της ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. 62 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 63 υπέρ. Α, όχι, όχι. Δεν ψηφίζουμε το ίδιο το 64, είναι ταυτόσημη 65. 65 υπέρ. Κατά απορρίπτεται 66 υπέρ κατά απορρίπτεται 67 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 68 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 69 υπέρ κατά απορρίπτεται. 70 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 71 ηλεκτρονικά. 71. Τροπολογία 71. Για το 71, κύριε Νταφ, προτείνω για την 71 να ψηφίσουμε δύο τμήματα ο ευρωσκεπτικισμός που αυξάνεται σε κάποια κράτη-μέλη, μέχρι εκεί το πρώτο τμήμα και το υπόλοιπο κομμάτι το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο που είναι το μόνο θεσμικό όργανο που ε, εκλέγεται άμεσα μέχρι τη λέξη citizens. Δύο λοιπόν τμήματα και ψηφίζουμε ξεχωριστά. Ψηφίζουμε λοιπόν το πρώτο τμήμα του 71 Το πρώτο τμήμα. Υπέρ. Υπέρ. Κατά. Α, ηλεκτρονικά καλύτερα να ψηφίσουμε. Αρχή της ψηφοφορίας για το πρώτο τμήμα της τροπολογίας 71. Τέλος. 13 υπέρ 13 κατά δεν εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα του 71. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Τέλος. Απορρίπτεται. 14 ε, κατά 12 υπέρ. Και τώρα περνάμε στην συμβιβαστική F. Ψηφίζουμε. Υπέρ κατά εγκρίνεται. 73. 73 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική G υπέρ κατά αποχές να επαληθεύσουμε καλύτερα. Αρχή της ψηφοφορίας, συμβιβαστική G. Πέρας. Εγκρίνεται. 14 υπέρ 11 κατά. Και τώρα ψηφίζουμε την 74-75 καταπίπτουν. Πάμε στην 79. 79 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεν υπάρχει μετάφραση από τα ουγγρικά στα ουγγρικά. 79, 79. Δεν υπήρχε μετάφραση στα ουγγρικά. Ψηφίζουμε λοιπόν τροπολογία του Ζωπιέρ Οντί. Υπέρ. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. 11 υπέρ, 11 κατά. Απορρίπτεται. 80 υπέρ κατά απορρίπτεται 81 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 82 δεν είναι παραδεκτή γιατί έχει να κάνει με μια διαδικασία η οποία αφορά τελικά την Επιτροπή Αναφορών. Δεν μπορούμε λοιπόν να την ψηφίσουμε, είναι μη παραδεκτή, 83 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, 84 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τελική τώρα ψηφοφορία την οποία θα κάνουμε ηλεκτρονικά. Άρχιτε ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με 22 ψήφους υπέρ, 4 ψήφους κατά, καμία αποχή. Ήταν πολύ κουραστική η ψηφοφορία βέβαια για όλους και προφανώς και για τους εισηγητές οι οποίοι όμως κατάφεραν τελικά να υποβάλουν ένα συμβαστικό κείμενο Υπήρχαν βέβαια και κάποιοι με επικεφαλή στην κυρία Λεγκρίπ οι οποίοι αντιτάχθηκαν σε κάποια σημεία και σας ευχαριστώ όλους πάντως για τη συνεργασία σας. Λοιπόν, περνάμε στην τελευταία ψηφοφορία για σήμερα.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 Είμαστε στο σημείο 8 της ημερησίας διάταξης. Έκθεση Επιτροπής για την επικουρικότητα και την αναλογικότητα. 19η έκθεση σχετικά με τη βελτίωση νομοθεσίας για το έτος 2011. 43 τροπολογίες έχουν κατατεθεί και να σας πω την αλήθεια δεν έχουμε καταφέρει καν να τις συζητήσουμε όλες. Γι' αυτό το λόγο δεν ξέρω αν κάποιος θέλει τώρα να πάρει το λόγο για να εξηγήσει συγκεκριμένες τροπολογίες. Κανείς όμως δεν θέλει να πάρει το λόγο από ό,τι βλέπω. Άρα μπορούμε να ψηφίσουμε Προτού όμως ξεκινήσουμε την ψηφοφορία, να σας πω εγώ κάποια πράγματα. Θα ήθελα να αποσύρω την δική μου τροπολογία, την υπαριθμών Sì, esatto. Quindi intendo ritirare il mio emendamento 27. 27. Αποσύρω την τροπολογία μου παριθμών 27. Μπορούμε τώρα να ψηφίσουμε. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με 14 υπέρ, 6 κατά. 4 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρτε ψηφοφορία. Πέρας. εγκρίνεται με 13 ψήφους υπέρ και 9 κατά. Τροπολογία 2 υπέρ κατά. Μα δεν σηκώνετε τα χέρια σας όμως, ηλεκτρονική ψηφοφορία για την τροπολογία 2, άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 18 υπέρ 6 κατά. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Με συγχωρείτε. Συμβαστική τροπολογία α υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 8 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 9 του κυρίου Ντάφ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία B υπέρ. Κατά. Κύριε Πρόεδρε, μπορούμε να έχουμε κατατμήματα όσον αφορά τις τρεις αυτές λέξεις all forms of. Γιατί δεν αληθεύει το ότι και όλες οι μορφές επηρεάζονται. Θα ήθελα λοιπόν να είχαμε χωριστή ψηφοφορία για τις τρεις αυτές λέξεις all forms of. Μα έχουν ήδη αποσυρθεί από το κείμενο οι λέξεις αυτές, λέει ο Πρόεδρος. Η συμβαστική τροπολογία δεν περιλαμβάνει τις τρεις αυτές λέξεις οποίες συνεφερθήκατε, άρα μπορούμε να ψηφίσουμε. Συμβαστική τροπολογία B υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Άρα μπορούμε να περάσουμε στην τροπολογία 15. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 16 τώρα. Ναι, πρέπει να την ψηφίσουμε, άρα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Με... Ναι, τροπολογία 16 απορρίπτεται, με συγχωρείτε λέει ο πρόεδρος. Τροπολογία 17 Κύριε Πρόεδρε, τι έγινε με τη 16. Λοιπόν, τροπολογία 16 του κύριου Νταφ. Η τροπολογία αυτή εγκρίθηκε. Συγγνώμη, μάλλον κουράστηκα, λέει ο Πρόεδρος. Να κάνουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Η γραμματεία μου λέει ότι δεν ήταν σαφές το αποτέλεσμα, άρα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για τροπολογία 16. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται για δύο ψήφους. Τροπολογία 17 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 22 22 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση για τροπολογία 22. Πέρας. Εκτός μικροφώνου. Νομίζω ότι έχει γίνει ένα λάθος στον κατάλογο ψηφοφορίας μας. Μας δίνετε λίγο χρόνο για να κάνουμε μια διόρθωση. Μα δεν έχει ολοκληρωθεί καν η ψηφοφορία. Λοιπόν, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την τροπολογία 22. Πέρας. Απορρίπτεται. 5 προς 19. Άρα μπορούμε να ψηφίσουμε τώρα τη συμβαστική C υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Άρα μπορούμε να περάσουμε στην 27, η οποία έχει αποσυρθεί. 25 λοιπόν και 26. Αυτές οι δύο είναι ταυτόσιμες, άρα τις ψηφίσουμε από κοινού, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. 28 Ψηφίζουμε την τροπολογία 28 του κύριου Ντάφη, υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται συμβαστική τροπολογία D υπέρ. Κατά. Αποχές. Συγγνώμη, νόμιζα ότι επρόκειτο για χωριστή ψηφοφορία σε δύο τμήματα. μέχρι το πρώτο κόλ. Ναι, όντως ψηφίζουμε λοιπόν κατά τμήματα. Ah, ecco. Sì, c'è una richiesta di parti separate da parte dei liberali, non era segnata quindi la mia Όντως ψηφίζουμε κατά τμήματα, πρώτο τμήμα, υπέρ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 6 προς 19. 43 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την 43 άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 17 υπέρ 8 κατά. Άρα καταπίπτουν οι τροπολογίες 39, 42, 40 και 41. Και μπορούμε να προχωρήσουμε στην τελική πλέον ψηφοφορία. Ψηφίσουμε ηλεκτρονικά το σύνολο του κειμένου, το σύνολο του ψηφίσματος. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. εγκρίνεται. 24 υπέρ, καμία ψήφος κατά και καμία αποχή. Ολοκληρώσαμε λοιπόν τις ψηφοφορίες μας. Και να σας πω ποιες είναι οι ημερομηνίε για τις επόμενες συνεδριάσεις. 5η 24 Οκτωβρίου στις 9 με 11 στο Στρασβούργο, έκτακτη συνεδρίαση. Τακτική τώρα συνεδρίαση θα γίνει στις 25 Νοεμβρίου από τις 3 ως 6.30 Βρυξέλλες. Σας υπενθυμίζω και κάτι ακόμα, ότι την 3η 26 Νοεμβρίου από τις 9 10 το πρωί θα διεξαχθεί σεμινάριο με τις μη ομολογιακές οργανώσεις και με τις εκκλησίες. Λύεται συνεδρίαση και στις 7 η ώρα έχουμε τη συνεδρίαση των συντονιστών. Μπορείτε να επαναλάβετε τις ημερομηνίες των συνεδριάσεων, δεν τις κατάλαβα. Αναφερθήκατε στην 24η Οκτωβρίου. Λοιπόν, ησυχία παρακαλώ, επαναλαμβάνω τις ημερομηνίες. 24 Οκτωβρίου από τις 9 ως 11 το πρωί συνεδριάζουμε εκτάκτως στο Στρασβούργο. Στις 25 Νοεμβρίου από τις 3 ως 6.30 το μεσημέρι συνεδριάζουμε στις Βρυξέλλες, τακτική συνεδρίαση. Και μετά στις 26 Νοεμβρίου από τις 9 το 10.30 το πρωί θα διοργανώσουμε αυτό το σεμινάριο που σας έλεγα προκειμένου να εφαρμόσουμε το άρθρο 17 της Συνθήκης της Λισαβόνας. Επομένως έχουμε ένα σεμινάριο με τις εκκλησίες και τις μη ομολογιακές ε, οργανώσεις λύεται η συνεδρίαση, αλλά στις 7 η ώρα θα έχουμε την συνεδρίαση των ιστών. Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη. Εφόσον ολοκληρώσαμε μισή ώρα νωρίτερα, Μήπω να ξεκινήσουμε και λίγο νωρίτερα, 7 παρατέταρτο, για παράδειγμα, τη συνεδρία των στονιστών. Με ευχαρίστω, λέει ο πρόεδρο. Αλλά δεν θα ήθελα να αποκλείσω κανένα από του τονιστές. Δεν ξέρω αν είναι όλοι ενήμεροι για το ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε νωρίτερα. κύριο Γκουαλτιέρη είπε να ξεκινήσουμε σε ένα τέταρτο. Εγώ θα μπορούσα ακόμα και τώρα να ξεκινήσω τι συνεδρία των συντονιστών. Η γραμματεία θα πάει να δει ποιοι είναι οι διαθέσιμοι παρόντες συντονιστές για να ξεκινήσουμε μια ώρα αρχίτερα.